Αξιότιμε ναι. κύριε πρόεδρε της Μογγολίας, αγαπητέ Έλμπερκτος, μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα που μπορούμε να σας καλωσορίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε πρόεδρε, η Μογγολία η πατρίδα σας, είναι ένα κράτος, μια χώρα με παλαιά και πλούσια πολιτιστική παράδοση, με ένα πληθυσμό, με μια δημοκρατία πολύ νεαρή και πολύ ζωντανή, παλόμενη δημοκρατία. Έγιναν το 1989 οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές. Πέρυσι εσείς ηγηθήκατε της ε, διαμόρφωσης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μπορέσατε μέσα από μια δύσκολη κατάσταση, να βοηθήσετε να βγει η χώρα σας, να έχει μια ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στεναρή. Η γεωγραφική θέση της χώρας σας μεταξύ των δύο μεγάλων και ισχυρών κρατών, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, είναι ασφαλώς δύσκολη μερικές φορές, το συζητήσαμε και στις δημιουργίες μας συνομιλίες, αλλά καθιστά ακόμη πιο εντυπωσιακά τα επιτεύγματα της Πολωνίας. Γιατί έτσι βλέπουμε πόσο ουσιαστική πολιτική μπορείτε να κάνετε και είναι φάρος στην περιοχή της η Μογγολία κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερω που μπορούμε να υποδεχθούμε σήμερα τον Πρόεδρο της χώρας, ο οποίος ε, θα είναι ο επόμενος οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής ΑΖΕΜ το 2016. Πρόκειται για μια σύνοδο πολύ σημαντική για την γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μια σύνοδο στην οποία περιφερειακά και διαπεριφερειακά προβλήματα μπορούν να βρουν λύσεις. Είμαι βέβαιος ότι μπορούν ε, οι συνομιλίε που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα τη χώρα σα να οδηγήσουν σε ουσιαστικέ λύσει. Και εμεί προσβλέπουμε και στην Συμφωνία Συνεργασία και Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μογγολία, που περιμένουμε να κυρωθεί από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Καλώ ήρθατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αξιότιμε κύριε Έλμπεντουρ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξοχότητες κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι απλό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε. Ευχαριστώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να συμμεριστώ τις απόψεις μου μαζί σας με σας τους ε, διακεκριμένους εκπροσώπους 28 κυρίαρχων κρατών αυτής της μεγάλης υπήρου της Ευρώπης. Είμαι ο νεότερος από 8 γιους. Για ε, πολλές γενιές ε, η οικογένειά μου ε, ζούσε ως νομάδες κτηνοτρόφοι στα δυτικά υψίπεδα της χώρας μου ε, στις βουνοκορφές Αλτάι. Οι γονείς μου ποτέ δεν είχαν ονειρευτεί ότι κάποια μέρα ο μικρότερος γιος τους θα μιλούσε από αυτό το έγκριτο βήμα προς ε, τις, εκείνες τις καρδιές στη δημοκρατία που ε, νοιάζονται ε, περισσότερο από κάθε άλλον για θέματα δημοκρατίας, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν πρόκειται για μένα. Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για το λαό μου και για τη χώρα μου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι περήφανος για την πατρίδα μου τη Μογγολία. Είμαι περήφανος για την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας και τη φυσική ομορφιά που μας περιβάλλει. Πάνω απ' όλα όμως είμαι περήφανος για το πνεύμα μας και για τις αξίες μας. Η σύντομη ιστορία της σύγχρονης ιστορίας του, της χώρας μου και το ταξίδι μας προς τη δημοκρατία θα ακουστεί οικείο σε πολλούς από εσάς. Στις αρχές της δεκαετίας του 20 η Μογγολία πέρασε υπό κομμουνιστική κυριαρχία η οποία διήρκεσε για 7 δεκαετίες. Κατά τις εκαθαρίσεις του Στάλιν ένας στους έξι ενήλικες σκοτώθηκε πάνω από 700 ναοί βουδιστικοί ε, κατακάηκαν. Οι ξένοι και εντόπιοι πράκτορες του κομμουνιστικού πειράματος στόχευσαν ακριβώς το πνεύμα του έθνους μου, αλλά δεν ήταν γραμμένο να κερδίσουν ούτε να διαρκέσει η κυριαρχία τους για πάντα. Στο τέλος κυριάρχησε η βούλησή μας να ζήσουμε ελεύθεροι. Μετά από πολλά χρόνια επιτέλους έφτασε η καθοριστική στιγμή για μας. Ένα κρύο πρωινό της 10 Δεκεμβρίου του 1989 οργανώσαμε την πρώτη δημόσια εκδήλωση στο δρόμο χωρίς έγκριση στην πρωτεύουσα Ουλαμπατόρ. Είχα την τύχη να εκλεγώ από τους συνοδοιπόρους δημοκράτες να συντονίσω εκείνη την ιστορική εκδήλωση. Μείναμε σιωπηλοί για πολύ καιρό. Τώρα είναι ώρα για δουλειά. Τώρα είναι ώρα για μεταρρυθμίσεις. Έτσι άρχισα την ομιλία μου τότε. Εκείνο το πρωινό απαιτήσαμε τα δικαιώματά μας, ελευθερία του συναθρίζεσθε, ελευθερία λόγου, ελευθερίας, ελευθερία του τύπου. Ζητήσαμε την δημιουργία ενός πολυκομματικού συστήματος, διεξαγωγή εκλογών και έναρξη μεταρρυθμίσεων στην αγορά. Ήταν η αρχή του ταξιδιού της χώρας μου προς την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και το άνοιγμα. Ήταν δύσκολο το ταξίδι που άρχισε. Εκείνη την εποχή γείτονη η Σοβιετική Ένωση ήταν ακόμα ανέπαφη και ο δραγμός, ο έλεγχός της ήταν ακόμα ισχυρός, σφιχτός ε, και κυριαρχικός. Στην πρωτεύουσα του άλλου γείτονα είχε γίνει σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν και το κρουστικό κύμα της ήταν ακόμα φρέσκο και ασκούσε επιρροή. Το παλιό καθεστώς ήταν επίμονο στη Μογγολία. Η παλιά νοοτροπία ανθίστατο στην αλλαγή. Οργανώσαμε πολλές εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, ε, απεργίας πείνας. Προσπαθήσαμε να ε, εξαλείψουμε κάθε λόγο για άσκηση βίας. Πάντοτε ζητούσαμε συμβιβαστικές λύσεις, ειρηνικές λύσεις. Και πραγματικά η δημοκρατική επανάσταση της Μογγολίας ήταν εντελώς ειρηνική. Δεν έπεσε ντουφεκιά, δεν έσπασε τζάμι, δεν άνοιξε μύτη. Σας ευχαριστώ. Ένα, σε ένα μήνα από τώρα η Μογγολία θα εορτάσει την 25η επέτειο ε, μετά τις πρώτες πολυκομματικές δημοκρατικές εκλογές. Από εκείνη την ιστορική ημέρα, στις 29 Ιουλίου του 1990, διεξήχθηκαν δημοκρατικές βουλευτικές εκλογές 7 φορές και προεδρικές εκλογές 6 φορές. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από 25 χρόνια, μετασχηματιστήκαμε από δικτατορία σε δημοκρατία. Παλαιά είμαστε ένα από τα πιο απομονωμένα κλειστά κομμουνιστικά καθεστώτα στον κόσμο και τώρα έχουμε γίνει ένα από τα πιο ανοιχτά καθεστώτα. Σήμερα έχουμε μια δυναμική οικονομία της αγοράς και μια σφίζουσα πολυκομματική, πλουραλιστική, δημιουργική κοινωνία. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ 20 Ο ιδιωτικός τομέας παράγει τώρα πάνω από το 80% του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένες αρετές που βρίσκονται στον πυρήνα της νεαρής μας δημοκρατίας. Αρετές που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε τα επόμενα χρόνια μέσα από τη συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και αλλού. Η ελευθερία του ατόμου είναι ο ακρογωνίος λίθος της δημοκρατίας μας. Οι Μογγόλοι αγαπούν την ελευθερία γιατί την κέρδισαν μέσα από σκληρή δουλειά. Η διακυβέρνηση, κυβέρνηση σε μια ελεύθερη χώρα δεν ε, είναι ιδιοκτησία μιας ομάδας ανθρώπων. Για να διατηρηθεί μια υγιής κοινωνία θα πρέπει να ε, ε καλλιεργείται και να αντιμετωπίζει προκλήσεις κάθε μέρα. Η ομορφιά της ελευθερίας είναι ότι είναι διαδικασία μάθησης. Είναι ένα σύστημα επούλωσης της ανθρώπινης κοινωνίας, ένα ε, σύστημα θεραπευτικό της κοινωνίας. Μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά δεν θα μας στοιχήσουν τη ζωή μας τα λάθη αυτά όπως γίνεται στις δικτατορίες. Γι' αυτό αγαπούμε την ελευθερία. Η Μογγολία είναι ανάμεσα στις ε, πρώτες ε, χώρες στον κόσμο ε, ανάλογα με τα ε, μέσα ενημέρωσης, ε, που, τα μέσα που χρησιμοποιούνται και τα εργαλεία των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά κεφαλή. Έχουμε τρία εκατομμύρια κατοίκους, αλλά είναι σαν να είναι και τρία εκατομμύρια δημοσιογράφοι παρόντες. Αυτό ως επιτοπλίστων είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει το δικαίωμα αμφισβήτησης της εξουσίας από το λαό και μας κάνουν ισχυρότερους η διαφάνεια και η αλληλεπίδραση. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που, είμαστε, ε, που προεδρεύουμε ε, στο συνασπισμό ε, της επιγραμμικής ελευθερίας. Καθώς η κοινωνία μας γίνεται πιο ανοιχτή, όλο και περισσότερο ακούμε ανήσυχες φωνές που ανησυχούν για την ασφάλεια. Όμως δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από τις καθολικές αξίες για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ασφάλειας του σήμερα. Βλέπουμε ότι συνεχίζει να εξελίσσεται και να απειλεί ο βίος εξτρεμισμός, αλλά η δέσμευσή μας σε αντίθεση υπέρ της δημοκρατίας, της ανεκτικότητας και της ειρήνης θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες. Γι' αυτό χαιρετίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξαιρετική πρωτοβουλία του να εγκρίνει έναν χάρτη θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων τον 21ο αιώνα. Ας συνεχίσουμε να εργαζόμεθα μαζί για να προωθήσουμε αυτή τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση. Δύο λόγια για τις εκλογές, την κυβέρνηση και τη λογοδοσία. Οι νέες τεχνολογίες ήταν ζωτική σημασίας για την υγεία της δημοκρατίας μας. Στις τελευταίες τρεις εκλογές χρησιμοποιήσαμε ηλεκτρονικά μηχανήματα για την ψηφοφορία και ένα βιομετρικό σύστημα καταγραφής των εκλογέων. Ε, αυτά είναι μέτρα που καταπολεμούν την απάτη και διασφαλίζουν στους εκλογείς ότι η συμμετοχή τους θα κάνει διαφορά. Βεβαίως η ε, ενστάλαξη της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση πάει πέρα από τις εκλογές. Οι Μογγόλοι ενδιαφέρονται στο πώς η κυβέρνηση δαπανά τα χρήματά τους που τα πληρώνουν μέσω των φόρων. Για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια έχουμε αναπτύξει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης. Ε, ο νόμος ε, για ε, την γυάλινη λογοδοσία που ε, επιτρέπει να, μια διάβγεια, ένα σύστημα σαν διά, τη διάβγεια που επιτρέπει να παρακολουθούν ε, τις δημόσιες δαπάνες ε, ηλεκτρονικά. Ε, η τεχνολογία έχει και την αντίθετη τάση. Γίνεται μικρότερη, πιο λειτουργική και πιο φιλική προς τους χρήστες ε, χρόνο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό ε, προχωρήσαμε σε μια έξυπνη πρωτοβουλία κυβερνητική η οποία ε, ενσωματώνει νέες τεχνολογίες ώστε η κυβέρνησή μας να μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες προκλήσεις. Η διαφθορά τώρα. Η διαφθορά είναι ένα μεταδοτικό νόσημα το οποίο αναπτύσσεται στο σκότος, καταστρέφει ε, κάθε θεμέλιο μιας ε, δίκαιης ε, και ασφαλούς κοινωνίας. Για να μπορέσουμε να κρυζώσουμε αυτό το κακό θα πρέπει να φωτίσουμε τη διαφθορά, να διασφαλίσουμε ότι θα την εκθέσουμε και θα εκθέσουμε και αυτούς που ευθύνονται για αυτήν που δεν πρέπει να ξεφύγουν από τη δικαιοσύνη. Είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια η Μογγολία ανέβηκε από το 120 στο 80 στον ε, δίκτυ ε, διαφθοράς της διεθνούς διαφάνειας. Ακόμα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά επιτελούμε πρόοδο σημαντική και καθαρίζουμε την αγαπημένη μας χώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ορισμένα άλλα ζητήματα. Θανατική ποινή και ανθρώπινα δικαιώματα. Κάναμε πρόοδο και στη σφαίρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το, το θεμέλιο της δικαιοσύνης είναι σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κεντρικό για, για την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Ε, επουδενή δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή η θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Πριν από, τον Ιούνιο, 18, ε, πριν από ε, τις 18 Ιουνίου 2009 η Μογγολία ε, βραβεύτηκε από την Διεθνή Αμνηστία ως μια ε, θεωρείται, συγγνώμη, συγχωρείτε, θεωρείτο από τη Διεθνή Αμνηστία ως ε, μια από τις χειρότερες χώρες σε ό,τι αφορά τη θανατική ποινή. Ε, ήταν τότε που ορκίστηκα πρόεδρος της Μογγολίας και την ίδια μέρα είχα δύο νομοσχέδια ε, στο γραφείο μου. Θα έπρεπε να ε, επιλέξω αν θα έπρεπε να επιτρέψω την εκτέλεση δύο ανθρώπων ή όχι. Επέλεξα τη ζωή. Επέμεινα στην απόφασή μου αυτή. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και άρχισα να περνώ αυτό το μήνυμα και στην κοινή γνώμη και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Δεν ήταν εύκολο να ασκήσω ε, τον ηγετικό μου ρόλο σε αυτό το θέμα, αλλά το 2012 η χώρα μου ε, επικύρωσε το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών που στόχο έχει την κατάργηση της θανατικής ποινής. Δεν έγιναν εκτελέσεις στη Μογγολία από τον Ιούνιο του 2009. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής πάνω σε αυτό. Η θανατική ποινή είναι αναποτελεσματική και βάρβαρη. Από αυτό το βήμα επιθυμώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους Ευρωπαίους φίλους που μας στηρίζουν και μας ενθαρρύνουν ε, σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Εξοχότητες, ε, η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος είναι επιτακτική για μας. Η μεταρρύθμιση του νομοθετικού και δικαστικού μας πλαισίου αποτελεί σημαντικό τμήμα των προσπαθειών μας οικοδόμησης μιας ελεύθερης και δίκαιης κοινωνίας. Ήταν μία από τις προτεραιότητές μου και κάναμε μεγάλα βήματα όλες τις πτυχές του δικαστικού συστήματος από την αστυνομία ε, στους ε, εισαγγελείς, δικαστήρια και δικαστές. Η εμπιστοσύνη του λαού ε, προς ε, ένα δίκαιο δικαστήριο αποκαταστάθηκε. Μια ελεύθερη κοινωνία θα πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς. Οι γυναίκες είναι η ραχοκοκαλιά της οικογένειας ε, και του έθνους. Φέρνουν τη ζωή στον κόσμο. Συχνά είναι εκείνες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των αρρώστων, όσων έχουν ανάγκη. Οι μητέρες μας, οι αδελφές μας, οι κόρες μας. Για να προχωρήσει μια κοινωνία χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες και στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο. I am proud to report... Είμαι περήφανος μπορώ να αναφέρω ότι κατά τις τελευταίες μας εκλογές τριπλασιάσαμε τον αριθμό των γυναικών στο κοινοβούλιο μας. Με περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας νομίζω ότι θα έχουμε μεγαλύτερη αρμονία, μεγαλύτερη συμμετοχή, λιγότερα προβλήματα και συγκρούσεις. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσης να πω Δύο λόγια για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, η παιδεία είναι η βάση για τη μελλοντική μας επιτυχία. Εγώ από μια οικογένεια ε, νομάδων κτηνοτρόφων έφτασα στο Χάρβαρντ. Κι άλλοι νέοι θέλουν να έχουν την ίδια ευκαιρία. Εργαζόμαστε σκληρά για να οικοδομήσουμε την ικανότητά μας στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες γιατί μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα για να ενισχύσουμε τα δικά μας ιδρύματα. Εξοχότητες, ε, κατα... αντιλαμβάνομαι ότι όλες οι δημοκρατίες όλες οι δημοκρατίες δεν πρέπει να είναι ίδιες. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις διαφορές. Η δημοκρατία είναι μια αντιπροσωπευτική μορφή ε, διακυβέρνησης. Σε κάθε έθνος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει ε, παραδόσεις και ε, κουλτούρα διαφορετική. Αλλά σε κάθε κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή περιορισμός της εξουσίας του κράτους, ε, να είναι δεκτικές οι κυβερνήσεις στα προβλήματα του κόσμου, να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να, επε, να, να στηρίζουν ε, υγιείς θεσμούς των πολιτών, να καταπολεμούν τη διαφθορά, να επιτρέπουν στον κόσμο να επιλέγει τους ηγέτες σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, αυτά είναι όλα θέματα όπου η Μογγολία και η Ευρώπη έχουν κοινέ αξίες και εδώ είναι που εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεργασία σας. Η Μογγολία και η Ευρώπη είναι παλιοί φίλοι, όπως καταδεικνύεται από μία επιστολή του Μογγόλου Κάνουλ Ζιτ προς τον Φίλιππο τον Ωραίο, ε, που εστάλει πριν από 710 χρόνια και λέει πώς μπορούμε να ε, λησμονήσουμε, για να επιτρέψουμε να λησμονηθεί η φιλία των προγόνων μας, των παππούδων, πατέρων και αδελφών μας που ε, αγαπούσαμε τόσο πολύ και που ενώ ήταν μακριά παρόλα αυτά ένιωθαν κοντά και αντάλλασαν λέξεις σοφίας και δώρα ειρήνης. Με το ίδιο πνεύμα σας μιλώ σήμερα ε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Μογγολίας-Ευρώπης. Ε, ε, με το τέλος, ε, την πτώση του κομμουνισμού, οι σχέσεις μεταξύ Μογγολίας και Ευρώπης άνθησαν ξανά. Η οικονομική, τεχνική, ανθρωπιστική σας βοήθεια και συνεργασία βοήθησε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας να οικοδομήσουμε μια ελεύθερη δημοκρατική κοινωνία και γι' αυτό είμαι θα ευγνώμονες Εξοχότητα το 2014 η Μογγολία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εόρτασαν την 25η επέτειο των διπλωματικών μας σχέσεων. Βλέπω τη συνεργασία με το ΞΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κράτους της Μογγολίας ε, ως κρίσιμο για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης. Ήδη έχουμε κάνει άλματα μπροστά συμπεριλαμβάνοντας την ε, θέσπιση της ε, Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ Μογγολίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τα κράτη-μέλη που επικύρωσαν τη συμφωνία. Και πράγματι υπάρχουν τώρα περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ για ευρωπαϊκές επενδύσεις. Ε, Πρώτη τάξης ευρωπαϊκές εταιρείε έρχονται στη Μογγολία για να επενδύσουν συχνά σε εταιρική σχέση με τις εταιρείε μας, σε συμπράξει. Ε, καθώς η κυβέρνηση παίρνει, κάνει βήματα για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, αυτές οι ευκαιρίες αυξάνονται ραγδαία. Ελπίζω ότι πολλοί από εσάς θα δείτε τις ομορφιές της χώρας μου και το δυναμικό που έχει από πρώτο χέρι το 2016 όταν η Μογγολία ε, θα είναι η περήφανη ε, χώρα που φιλοξενεί την ενδέκατη συνάντηση Ασίας-Ευρώπης. Ε, πραγματικά προσβλέπω να στο καλωσόρισμα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στη χώρα μου και σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι μια αξιομνημόνευτη σύνοδος. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η δέσμευση της Μογγολίας υπέρ της διεθνούς συνεργασίας είναι ισχυρή. Πρόσφατα ε, αρχίσαμε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται το βήμα της Ασίας. Ελπίζομαι ότι θα αποτελέσει ένα μηχανισμό που τόσο χρειαζόμαστε για να προωθήσουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση σε όλα τα κυρίαρχα κράτη της Ασίας, προωθώντας ίση εκπροσώπηση των διαφορετικών συμφερόντων τους. Η κυβέρνησή μου εργάζεται τώρα για να ολοκληρώσει αυτή την προσέγγιση και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν με ιδέες που θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Φίλοι μου, η Μογγολία δεν έχει καμία πρόθεση να δώσει μαθήματα σε κανέναν για τη δημοκρατία. Όμως έχουμε πολλά διδάγματα να μοιραστούμε. Με το Κυργιστάν ε, μοιραζόμεθα τα διδάγματα που αποκομίσαμε ε, οικοδομώντας αποτελεσματική ε, κοινοβουλευτική δημοκρατία και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Με το Αφγανιστάν ε, διοργανώνουμε εκπαίδευση για διαδιπλωμάτες και δημοσίους υπαλλήλους. Με την Μιανμάρ κάνουμε εκδηλώσεις για δημοσιογράφους, μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Με τη Βόρεια Κορέα ε, διεξάγουμε οικονομικό διάλογο και διάλογο για την ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι η Μογγολία μπορεί να συμβάλλει πολύ σημαντικά στην περιφερειακή ασφάλεια στη Βορειοανατολική Ασία και πέραν αυτή. Καταλαβαίνουμε τις ε, επιπτώσεις του ψυχρού πολέμου. Λόγω της εμπειρία μας ε, και επί και επί δημοκρατίας έχουμε την μοναδική δυνατότητα να παίξουμε το ρόλο ενός έντιμου διαμεσολαβητή υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή μας το, το 2013 ε, ανακοίνωσα το διάλογο του Λαν ε, για την ασφάλεια στην Βορειοανατολική Ασία. Επίσης φιλοξενήσαμε μία σειρά από συναντήσεις και διασκέψεις ε, επιθεμάτων πέρα από την ασφάλεια όπως ενέργεια, γυναίκες, πυρηνικά θέματα. Η χώρα μου ζητούσε, ε, επιζητούσε επί 23 χρόνια να αποκτήσει καθεστώς ελεύθερο πυρηνικών. Το 2012 τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπέγραψαν μια κοινή ε, δήλωση ε, επιβεβαιώνοντας ε, το καθεστώς μας ελεύθερο πυρηνικών. Οι Μογγόλοι λένε ο καλύτερος άνθρωπος δοκιμάζεται στην ανάγκη. Το καλύτερο άλογο δοκιμάζεται στην υπασία. ε, έσπευσα να διαβάσω μια σελίδα ε, μετά. Επανέρχομαι. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ενώ η πυρηνική σχέση μπορεί να παραμείνει βιώσιμη για κάποια χρόνια, οποιοδήποτε έθνος ε, επιδιώκει να δημιουργήσει πυρηνικά δεν πρέπει να ε, υπονομεύει την ειρήνη και την ασφάλεια των γειτόνων, τους, των γειτόνων του. Εμείς ε, αναλαμβάνουμε την ευθύνη πολύ σοβαρά για την προώθηση της ειρήνης. Οι, οι ένοπλες δυνάμεις της Μογγολίας ε, φορούν με περηφάνεια ε, του, ε, το, το κιανό κράνος και έχουμε συμβάλει επί ε, στην ειρήνη μαζί ε, με άλλους 20 μεγάλους ε, που εργάζονται για την ειρήνη. Εμείς είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε υπηρεσίες και συμβάλλουμε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και τα έθνη τη Ευρώπη, διότι συνεχώ υποστηρίζετε τη χώρα μου, τη Μογγολία. Οι Μογγόλοι λένε ο καλύτερος άνθρωπος δοκιμάζεται στην ανάγκη και το καλύτερο άλογο δοκιμάζεται στην υπασία. Είσαστε μαζί μας όταν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας πάρα πολύ. Είσαστε μαζί μας όταν χρειαστήκαμε τη φωνή σας για να μας ενθαρρύνει. Είσαστε πάντοτε με τη Μογγολία και μας ενθαρρύνατε και μας επιβραβεύατε ε, στις επιτυχίες μας και μας βοηθούσατε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ε, μοναδική για την προώθηση της ευημερίας σε όλο τον κόσμο, την προώθηση της ειρήνης και της αρμονίας. Η Μογγολία θα είναι στρατηγική άγκυρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ανατολή θα βοηθήσει να προχωρήσουμε τις κοινέ μας αξίες και συμφέροντα για να οικοδομήσουμε την ειρήνη, τη δημοκρατία και τη συνεργασία στην Ασία. Φίλοι, ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. meine sehr geehrten Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι ομιλώ εκ μέρου όλων σα ευχαριστώντας τον Πρόεδρο για την ομιλία του, έστω και αν πέρασε μια σελίδα από λάθο. Πρέπει να πω ότι και πάλι εκ μέρου όλων των συναδελφών ότι χρόνια τώρα δεν είχαμε ακούσει τόσο ε, αισιόδοξο μήνυμα, τόσο ενθαρρυντικά λόγια και εμείς υποστηρίζουμε βεβαίως και σας ευχαριστούμε για την ένθερμη υποστήριξη συνεργασίας της χώρας σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε.